Να αρχίσουμε συνάδελφοι, λέει πρόεδρος. Πρώτα πρώτα όμως έχουμε ένα διαδικαστικό, το οποίο προέρχεται από τον κύριο Μόλτσε. Κυρία Πρόεδρε, άρθρο 145 του κανονισμού στις 24 Απριλίου ο Χάντς Πέτερ Μάρτιν εν απουσία μου κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών υποστήριξε ότι από τη θέση μου έγινε κάποια ψηφοφορία με κάρτα. Βεβαίω το Προεδρείο είπε ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό Καταλαβαίνω βεβαίω ότι εν των εκλογών κάποιοι συνάδελφοι βρίσκονται σε μια ειδική ε, ψυχολογική κατάσταση. Αλλά το να κατηγορείται κάποιο ω απαταιώνα ότι ή ότι δέχεται να γίνεται κάποια πάτη στο όνομά του είναι υπερβολικό. Πιστεύω ότι. Ε, δεν, ε, ότι πρέπει να διαμαρτυρηθώ και ξέρουμε πολύ καλά ότι ε, και άλλες φορές ε, ε, με έχει κατηγορήσει ο συνάδελφος για πολλά πράγματα έφτασε τώρα στο τώρα είμαστε εκτός πραγματικότητας νομίζω υπερβολικά τα πράγματα οπότε ζητώ να αποσύρει αυτά που είπε Ευχαριστώ κύριε Μόλι, όπως γνωρίζετε έγινε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε κάποια, κάποιο πρόβλημα, κάποια χειραγώγηση της χρήσης της συσκευή. Τέλος πάντων, ο Γιώργος Χάνης Πέτερ Μαρτίν θέλει τον ε, λόγο. Παρακαλώ να είστε σύντομος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα να σας ζητήσω να, γίνει γίνει μια κάποια ησυχία ή τελικά μένα προσπαθείτε να τιμωρήσετε. Εκατόν σαράντα είναι το άρθρο ε, για την προσωπική παρουσία παρατήρηση που έκανε ο συνάδελφος ζητήθηκε να ζητήθηκε να ε, αποσύρω ορισμένα πράγματα που είπα για τους εξτρεμιστές της δεξιάς και τα λοιπά ε, όντως είπα εγώ κάποια τέτοια πράγματα και ακούτε και κραυγές εδώ οι οποίες δείχνουν ακριβώς ότι δίκιο έχω με την ε, καταγγελία αυτή για εξτρεμισμό της δεξιάς πραγματικά στο παρελθόν πολλές φορές ελέγξαν πολλά κακά πράγματα εναντίον μου αλλά οι... δεν έχουν λόγο ύπαρξης καταγγελίες αυτές διότι οι δικαστές της Αυστρίας θα είχαν ασχοληθεί με την περίπτωσή μου εάν υπήρχε και ένας κόκκος αλήθειας μα έχει ευκαινιστεί το θέμα αρκεί τώρα λέει η κυρία για, να αρχίσουμε τώρα. Έχουμε βέβαια και άλλο ένα διαδικαστήριο. Κύριε Ντονίτσι, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, αλλά δεν το γνωρίζουν πολλοί συνάδελφοι, λόγω της ε, λοιπούς ε, ενημέρωσης που δίνεται από το Προεδρείο για αυτή την υπόθεση που θέλουμε να περάσει σιωπηρά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε για την ε, μακρά διαμάχη την οποία, η οποία με, έχει φέρει σε αντίθεση με τον κύριο Κέτο εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο. Στις 24 Μαρτίου δεν επικυρώθηκε η δική μου εντολή λόγω της ε, καταγγελίας των Εθνικών Αρχών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάστηκε να καταβάλει τις δαπάνες. Η, απόφαση του δικαστηρίου είναι η αποκατάσταση της θεμητής, ε, της νόμιμης μάλλον ε, διαδικασίας του Κοινοβουλίου. Αντίθετα, ο πρόεδρος Πέτερινγκ στις 17 Μαΐου έδωσε μία αμφίβολη θέση προβαίνοντας στην επαλήθευση των δικών μου ε, διαπιστευτηρίων και όχι μόνο αυτό, αλλά συγκάλεσε έκτακτα την Επιτροπή και επειδή αυτή είναι η τελευταία ολομέλεια της θητείας, εκτός και αν παραταθεί η δική μου εντολή και στην επόμενη θητεία, θα ήθελα να καλέσω την Προεδρία να διορθώσει αυτή την, αυτό το περαιτέρω χονδροειδές σφάλμα ε, και να συμφωνήσει με την απόφαση του ΔΕΚ. Θα ήθελα να μην είχε γίνει όλη αυτή η νομική ήττα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ωστόσο θα ήθελα να σας χαιρετήσω με μεγάλη εγκαρδιότητα σας προσωπικά. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τόνιτς, τα σχόλιά σας έχουν καταγραφεί και φυσικά ο Πρόεδρος ε, προέβησε δήλωση τη Δευτέρα το απόγευμα και τα σχόλιά σας θα διαβιβαστούν στο απόψινό, στην απόψινή συνεδρία του Προεδρείου. Επόμενο θέμα είναι η ψηφοφορία για την πρόταση απόφασης για τις ε, αρμοδιότητες και ευθύνε. Και έχουμε την πρώτη τροπολογία και θα την ψηφίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Όχι, δεν σαφέ το αποτέλεσμα. Πρέπει να γίνει έλεγχος, ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε, ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε το σύνολο της απόφασης με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το επόμενο θέμα αφορά το σχέδιο απόφασης όσον αφορά τις δικοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες. Κύριε Βίρτ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πολιτική μας ομάδα θα ήθελε να γίνει χωριστή ψηφοφορία όσον αφορά την παράγραφο 1 εδάφιο α και σας ε, ονομάζω εκεί που λέει η αντιπροσωπεία με τις σχέσεις με Αλβανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο και Πέδιο. Διότι κατά τη γνώμη μας ε, εδώ de facto αναγνωρίζουμε το Κόσοβο, κάτι το οποίο είναι απαραίδεκτο. Παρακαλούμε αυτή η παράγραφος να περάσει από χωριστή ψηφοφορία. Είναι εκπρόθεσμα το αίτημα, αλλά ε, εντάξει, αν δεν υπάρχει καμία ένσταση από ό,τι φαίνεται. Κύριε Πόσελ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, έχω σοβαρές ενστάσεις. Με τρία τέταρτα ε, πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την ανεξαρτησία του κοσφοπεδίου. Το βρίσκω απαράδεκτο να αμφισβητείτε τώρα. Πρόεδρος, συμφωνείτε να γίνει χωριστή ψηφοφορία ή θα πρέπει να ψηφίσουμε από αυτό. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένσταση σε αυτό το αίτημα. Επομένω θα συνεχίσουμε όπως αρχικά προβλεπόταν. Πρώτη τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ της πρώτης τροπολογίας κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο του σχεδίου απόφασης με ονομαστική ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας εγκρίνεται το επόμενο αφορά την έκθεση μοριών σε σχέση με την οδηγία 83-515 και 11 αποφάσεων σαν την κοινή αλληλευτική πολιτική. Θα ψηφίσουμε όλες με τις διατάξεις, με ονομαστική, τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνονται. Συγχαρητήρια, κύριε Μοριγιό. Τα επόμενα. και πάλι του κυρίου Μοριών σε την κατάργηση 14 κανονισμών για την κοινή ελευθερική πολιτική. Μία και μόνη ψηφοφορία, ονομαστική, τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια και πάλι κύριε Σιγητά. Το επόμενο είναι Ε, στήριξη ερωτικής ανάπτυξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Ερωτικής ανάπτυξη με νοστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Το επόμενο. Έκθεση ονεστά για τη διαδικασία αναφορών. Ονομαστική ψηφοφορία. Απαιτείται ειδική πλειοψηφία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Ωνιστά. Το επόμενο είναι η έκθεση Μπέγκε όσον αφορά την τροπή της Διοργανικής Συμφωνίας για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο ψηφίζουμε ονομαστική ψηφοφορία και πάλι χρειάζεται και εδώ ειδική πλειοψηφία ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια εισηγητά. Το επόμενο. Έκθεση Haug. Σχέδιο διορθικού προπολογισμού. Για τη χρήση του 2009 και εδώ χρειάζεται δική πλειοψηφία, ονομαστική. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το επόμενο. Έκθεση Χάου όσον αφορά διορθωτικό συμπληρωματικό προπολογισμό για τη χρήση 2009 και πάλι ονομαστική ψηφοφορία Ειδική πλειοψηφία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. κρίνετε συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Το επόμενο είναι πρόταση ψηφίσματος. Πρόκειται από την Επιτροπή Βιομηχανίας όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας των τηλεράσεων. Κραστική πλειοψηφία, δεν έχουμε τροπολογίε. Ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Το επόμενο. Πρόταση ψηφίσματος. Επιτροπή Βιομηχανίας όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας των οικιακών ψυχτικών συσκευών και πάλι ειδική πλειοψηφία και ονομαστική. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτωτο. Διότι δεν συγκέντρωσε την ειδική πλειοψηφία. Πρόταση ψηφίσματος. Επιτροπή Ανάπτυξης πρόγραμμα δράσης 2009. Μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές για ανάπτυξη. Απλή πλειοψηφία απαιτείται, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το επόμενο. Έκθεση Κόρμπετ. Γενική αναθεώρηση του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Έχουμε το από την Αρμαδία Επιτροπή. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές, εγκρίνεται. και τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία υπαριθμών 9 με χωριστή ψηφοφορία σε τρία τμήματα. Ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Και αυτό με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέραστη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Κυρία Φρασόνη, δείτε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ενημερώσαμε τις υπηρεσίες σε σχέση με την αναπομπή στην Επιτροπή. Αλλά δεν είπατε τίποτα και αρχίσατε την ψηφοφορία. Όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ήξερα τίποτα γι' αυτό, λέει η Πρόεδρος. Ναι, το ζητήσαμε, λέει η κυρία Φρασόνη. You can make the request. Μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημα, λέει η Πρόεδρος. Παρντών, λέει η κυρία Φρασόνη. Δυνάμει του άρθρου 168 μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημα ανα πάσα στιγμή μέχρι την τελική ψηφοφορία. Καλά, λέει η κυρία Φρασόνη. Τότε υποβάλλω το αίτημα να μπει στην Επιτροπή και να σας εξηγήσω το γιατί. Thank you very much, uh, President. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε κατά κοινοβουλευτική θητεία έγινε πολλή συζήτηση όσον αφορά τη μερίδα των επιπτώσεων, δηλαδή κάθε φορά που θεσπίζεται ένας νέος ε, κανόνας θα πρέπει κανείς να εξηγήσει ποιες είναι οι επιπτώσεις. Για δε τον νέο κανονισμό που θα ψηφίσουμε σήμερα βάσει της έκθεσης Κόρμπετ δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Αυτή της ε, εκβάθρων διότι θα είναι δυνατόν να έχουμε κοινέ επιτροπές πολλούς συντάκτες στην Ολομέλεια, στην τελική ψηφοφορία όπου θα έχουμε αντίφαση στις ε, διαδικασίες αλλά και στις τροπολογίες και για αυτό η παραταξή μας ζητεί να αναπαινθεί το κείμενο στην Επιτροπή όχι γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση αλλά διότι θεωρούμε ότι αν προχωρήσει αυτή η μεταρρύθμιση η δουλειά στο κοινοβούλιο θα γίνει πολύ δύσκολη. Κυρία Φασόν, σας ευχαριστώ και τώρα. Ένας αγορητής κατά. Αλλά ο εισηγητής κύριε Λάινεν, θέλετε να μιλήσετε κατά. Ναι κυρία Πρόεδρε, Ευχαριστώ. Η μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ δύσκολη. Ε, φαίνεται όμως ότι η μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ακόμη πιο δύσκολη. Λέει η κυρία Μισό φρασώνει ότι δεν είναι ε, καλές οι αλλαγές που έγιναν μέχρι τώρα αλλά έλαβε εκείνη μέρος στην όλη μεταρρύθμιση που γίνεται εδώ και δυόμισα χρόνια έγιναν πολλές συζητήσεις πάρτηκαν πολλές αποφάσεις σε αυτά τα δυόμιση χρόνια δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναπέμψουμε το θέμα στην Επιτροπή επιτέλους θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα έχουμε καιρό να ε, κάνουμε κάτι καινούριο αν θέλουμε στην επόμενη θητεία. Κατά λοιπόν τη κυρία ε, κυρίας Φρασόνη. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα κυρία Πρόεδρε εκτό του ότι η αιτιολόγηση εκ μέρους της κυρίας Φρασόνη ίσως είναι λόγο εκείνη να καταψηφίσει αυτέ τι τροπολογίε. Σίγουρα όμω, δεν αρκεί αυτή, αυτή, αυτή, η λόγια αναπομπή του συνόλου του κειμένου και έτσι να μην ψηφίσουμε τίποτα. Νομίζω ότι η πρόταση είναι ατύχης. Ψηφίζουμε, λέει ο πρόεδρος. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης Φρασόνη να γίνει αναπομπή στην Επιτροπή. Thank you. Ποιοι είναι κατά της πρότασης Φρασόνη. Αποχές. Είναι σαφές το αποτέλεσμα. Θα συνεχιστεί η ψηφοφορία. Ήμασταν στο τρίτο τμήμα της τροπολογίας 9 για μια ονομαστική ψηφοφορία και ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Τέλος της εφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11, ονομαστική. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 23. Έχω στην ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 29 χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 Χωστή ψηφορία. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για το 32. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται και πάμε στο 33 με χωριστή ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Ονομαστική. Ονομαστική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα του 33. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. 33. Ονομαστική. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτω ότι δεν συγκεντρώθηκε η απαραίτητη δική πλειοψηφία και πάμε στο 42 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. And that is adopted. Εγκρίνεται πάμε στο 45. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να γίνει έλεγχος επί του 45. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το Τροπολογία 51. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62. Ονομαστική. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Χωριστή ψηφοφορία. Ονομαστική. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα για το δεύτερο τμήμα της ε, τροπολογίας 8. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 61 η οποία έχει αποσυρθεί. 63 με ονομαστική. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται και πάμε τώρα στο 10 με ονομαστική. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Δεν Εγκρίνεται. 53. Μια ονομαστική. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 14. Υπέρα κατά αποχές εγκρίνεται Ναι, να γίνει έλεγχος γιατί χρειάζεται δική πλειοψηφία. Ψηφίζουμε το 14. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεν Υπάρχει μια συμβιβαστική τροπολογία. Η 69. Δυναμή το άρθρο 154 του κανονισμού απαιτείται να συμφωνήσει το σώμα πριν η τροπολογία αυτή ψηφιστεί. Έχει κανείς αντίρρηση. Όχι. Άρα, έχουμε τη συμβαστική για το 69. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ να κάνουμε έλεγχο για το 69. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Απολογία 17, χωριστή ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Το πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορείτε γιατί απαιτεί το ειδική πλειοψηφία, αλλά αν θέλετε να κάνουμε έλεγχο. Δεύτερο τμήμα. Υπό. Υπέρ, ποιο είναι, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 59. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. άποχέ. Εγκρίνεται. 64. Με ονομαστική. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54 μας και ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτωται, 57 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτωται. Ο κύριος Κόρμπετ ζητεί το λόγο. Πρόεδρε, πριν ψηφίσουμε το 49 και το 67, παρακαλώ αντιστρέψτε τη σειρά να ψηφίσουμε πρώτα το 67. Διότι έτσι στην Επιτροπή την Κοινοβουλευτική διαμορφώθηκε ο συμβασμό και γι' αυτό είναι η λογική τη των πραγμάτων. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση αφού εσεί το προτείνετε που είστε ο συγητή. Οπότε πρώτα να ψηφίσουμε το 67 με ονομαστική ψηφοφορία, λέει πρόεδρο. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτοντα και ξαναγυρίζουμε στο 49 ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε Ψήφισαν όλοι. Ξέρετε πώς να ψηφίσετε. Ξέρετε τι ψηφίζετε. Ωραία, είχατε χρόνο να το σκεφτείτε καλά και τώρα τέλειωσε η ψηφοφορία και εγκρίνεται. Άρα απορρίπτεται το 65. Οπότε τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου της αποφάσεως με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Κύριε Κόρμπετ. Τώρα όμως θα γίνει μια διακοπή εις τις ψηφοφορίες.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, σε μερικές εβδομάδες μεταξύ και 7 Ιουνίου οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκλέξουν